Κυρίες Κυρίε και κύριοι, ασφαλώ έχετε ενημερωθεί όλοι για την ε, σοβαρή υπόθεση του σοβαρού επεισόδιο που έλαβε χώρα εδώ. Ο συνάδελφο Παπαστάμκος πέρασε ένα σοβαρό ιατρικού χαρακτήρα επεισόδιο. Δεν είμαι σε θέση να σας ενημερώσω για την οριστική διάγνωση. Αλλά η κατάσταση είναι σοβαρή. Οι συνάδελφοι οι οποίοι ε, φρόντισαν πρώτοι τον κύριο Παπαστάμκο εδώ ε, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, τον κύριο Τάνοκ, τον κύριο Ζουλβέρ, την κυρία Κόμη ιδιαιτέρως εσάς που πρώτοι προσέφεραν τις βοήθειες στον κύριο Παπαστάμκο αυθόρμητα σε μια κατάσταση ασυνηθίστε. Και ελπίζω ότι βοηθήσατε τον κύριο Παπαστάμκο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπαστάμκος Ο κύριος Παπαστάμκος είναι τώρα στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να πω τίποτε το οριστικό για τη διάγνωση όπως σας είπα. Μόλις ενημερωθούμε από το νοσοκομείο για τη διάγνωση θα σας την κοινοποιήσω. Για το τι πρόκειται, για το τι πρόβλημα υπάρχει, για το τι ε, διάγνωση υπάρχει και φυσικά αυτό με κάθε σεβασμό της, ε, του απορρίτου του ιατρικού. Πάντως η κατάστασή του είναι σοβαρή, αυτό πρέπει να σας ε, πω. Έχω ενημερώσει την οικογένειά του, η σύζυγός του βρίσκεται στον δρόμο του Στρασβούργου. Είναι πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι αιτιολογημένα πιστεύω μου ζήτησαν να μην ε, προχωρήσουμε στις ε, ψηφοφορίες αυτή τη στιγμή. Δεν ήθελα να σας επισημάνω. ότι δεν μπορούμε να ξανακάνουμε ογκοδέστατες ψηφοφορίες σαν αυτή που είχαμε σήμερα. Εγώ είχα απορρίψει την πρόταση αυτή. Διότι θεώρησα ότι είναι υπερβολική. Αλλά η Επιτροπή δεν μπόρεσε να περιορίσει τον αριθμό των πολλών τροπολογιών. Και πρέπει να πω εδώ ότι όλες οι ομάδες μου είχαν επισημάνει ότι επιθυμούσαν τη διεξαγωγή αυτής της ε, ψηφοφορίας. Ένας συναδέλφος ζήτησε σήμερα την αναβολή της ψηφοφορίας. Απερίφθη η πρόταση. Αυτό ε, μας υποχρεώνει όλους να ξανασκεφτούμε πολύ σοβαρά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι κάποιος είναι υπεύθυνο ή υπέτειος, πρέπει να αναζητήσουμε άλλους τρόπους ώστε να μην χρειαστεί να ψηφίζουμε για τελείωτες ώρες. Όταν πια μάλιστα στο τέλος της ούτε καν γνωρίζουμε τι έχει ψηφίσει ο καθένας, ποια είναι η κατεύθυνση της πληροφορίας, γιατί είναι δύσκολο να έχουμε μια εικόνα συνολική. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους συναδέλφους να συζητήσουμε στη διάσκεψη των Προέδρων μια διαφορετική λύση. Πάντως πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα αυτού του περιστατικού και να αναλογιστούμε αυτή την υπόθεση. Παρακαλώ λοιπόν όσοι μπορούν να προσευχηθούν να προσευχηθούν, όσοι μπορούν να ελπίσουν να ελπίζουν, να δούμε τον κύριο Παστάμκο σύντομα κοντά μας, κοντά μας υγιή, γερό και δυνατό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίσιμες οι ώρες και όλοι πράγματι προσευχόμαστε για τον κύριο Παπαστάμκο επειδή όμω αναφέρθηκε και ο πρόεδρο Σούλτ στο τι συνέβη και γιατί είχαμε μακρά ψηφοφορία κτλ., θα ήθελα να παρακαλέσω το Προεδρείο σα να εξετάσει τι ακριβώ συνέβη και για πάρα πολλή ώρα, όπω ο ίδιο ο πρόεδρο ανέφερε, οι συνάδελφοι, οι ιατροί συνάδελφοι ήταν εκείνοι που φρόντιζαν τον Παπαστάμκο και όχι αυτοί που θα έπρεπε. Και πολλοί άργησαν να έρθουν στην ώρα του επάνω από τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου μα για να προσφέρουν τι πρώτε βοήθειε. Παρακαλώ να ερευνηθεί αυτό, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι βέβαια, όλων μας οι σκέψεις ε, είναι στον κύριο Παπαστάμκο. Ο κύριο Σούλτ όμω, ε, για να αναφέρω ένα άλλο θέμα, μα ε, κάνει υποδείξει το πώ θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μα. Εγώ θα υπερασπιστώ το έργο τη Επιτροπή Γεωργία και θα πω ότι ξέρουμε πώ πρέπει να γίνεται η δουλειά μα. Ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου είπε ότι ψηφίζουμε για πράγματα και δεν γνωρίζουμε προ ποια κατεύθυνση ψηφίζουμε. Α είμαστε ειλικρινεί, τουλάχιστον το λέω εγώ προσωπικώ για το δικό μου γραφείο. Δεν μπορούμε να έχουμε προσωπικό που δουλεύει 24 ε, ώρε το 24ωρο. Αυτό συμβαίνει εδώ. Είναι υπερβολική η πίεση, ο όγκο των εκθέσεων που μας αναλογή. Και ίσω θα πρέπει αυτό να κοιτάξει ο πρόεδρο Σούλτ. να κάτσουμε κάτω και να βρούμε καλύτερου τρόπου εργασία. Ο όγκο, το υλικό που έχουμε να χειριστούμε και να μελετήσουμε, δεν είναι δυνατόν να το χειριστούμε και να το μελετήσουμε κατά τρόπο αποτελεσματικό. Έκανε θαύματα η Επιτροπή τη γεωργία για να περιορίσει τι 8.000 τροπολογίε σε κάποιο έγγραφο σχετικά συνεπές και συνεκτικό. Η δημοκρατία αυτό μας καλεί να κάνουμε, να επιτρέπουμε στους ε, βουλευτές να ψηφίζουν τις προτάσεις. Αυτό ήταν και το νόημα της σημερινής ψηφοφορίας. Ίσως λοιπόν να πρέπει να δαχθούμε, όπως είπε ο Πρόεδρος, από τα όσα είδαμε. Ας αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία ή μη τι άλλο να συζητήσουμε τον τρόπο εργασίας μας. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλοί ζητούν το λόγο. Για το τραγικό αυτό περιστατικό φαντάζομαι. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ο οποίος όπως και οι άλλοι και οι ιατροί που έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο ήταν παρόντες αμέσως εδώ το ιατρικό προσωπικό και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους συνεργάτες, βουλευτές όσοι ήταν εδώ και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Δεν είναι νομίζω η στιγμή τώρα. Εδώ στην Ολομέλεια και ενώ δεν γνωρίζουμε ποια είναι η έκβαση αυτής της υπόθεσης. Να αναλύουμε, να υπεραμεινόμεθα κτλ. Μια συζητήσεως. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου είπε, το εννοήσε, ήμασταν όλοι παρόντες, ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα αίτια και τις συνέπειες με ηρεμία, χωρίς να καταγγέλει κανέναν. Είπε ότι πρέπει να αναλογιστούμε και παρακαλώ να μην γίνει τώρα αυτή η συζήτηση. Να αφήσουμε να παρέλθει λίγος χρόνος ο Πρόεδρος ανέλαβε μόνος του την ευθύνη να συνεχίσει την ανάλυση και να διατυπώσει συμπεράσματα και να σας ενημερώνει διαρκώς για τις εξελίξεις. Σας παρακαλώ θερμά να μην συνεχιστεί τώρα αυτή η συζήτηση. Όποιος εξάπαντος του επιθυμεί φυσικά θα λάβει το λόγο. Δεν μπορώ να ε, υποχρώσω κανένα σιγά σιγά, αλλά παρακαλώ να μην παρασυρθούμε από την δύσκολη αυτή κατάσταση και να αφήσουμε να περάσει λίγο χρόνο να συστήσουμε το θέμα με πιο πολύ απόσταση και πάλι κάθε τις καλύτερες ευχές μας για τον φίλο κύριο Παπαστάμουκο. Κύριε Αγγέλο. Κύριε Πρόεδρε, στα όσα είπατε κι εσείς. Ύστερα από ένα περιστατικό όπως το παρόν δεν είναι η ώρα νομίζω να κάνουμε αναλύσεις απευθείας ή να κοιτάμε ποιος βρισκόταν πού, σε ποια χρονική στιγμή. Αλλά διαρωτώ αν μπορούμε να περάσουμε πάλι στη μέρη σε διάταξη. Τόσα όσα συνέβησαν σήμερα προκύπτουν ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, πραγμάτων που δεν λειτουργούν σωστά στο Κοινοβούλιο και ίσως αυτό θα ήταν ένας ε, τρόπος, μία μέθοδος να το καταγράψουμε. τουλάχιστον λοιπόν για σε ένδειξη και σεβασμό και της ε, μέρημνάς μας για τον κύριο Παστάμκο να μην συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την εβδομάδα και να μην ξαναβρεθούμε αύριο σε μια κατάσταση όπου καθένας από εμά διαπιστώνει ότι επί δυόμιση ώρες πατούσε ένα κουμπί. Γι' αυτό παρακαλώ το Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή, υπ' αυτές τις συνθήκες, για αυτή την εβδομάδα, να πούμε φτάνει. Κύριε